Andiamo. Good afternoon. Dear members. Χαίρετε, αγαπητά μέλη και αγαπητοί συνάδελφοι. Dear colleagues, dear members, please take your seat. Καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Αρχίζουμε σιγά σιγά. Thank you. Thank Καλώς ορίσατε όλοι σε αυτή τη μεικτή συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι για πρώτη φορά εφαρμόζουμε το άρθρο 51 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Το άρθρο 51 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπαμε, μας δίδει την ευκαιρία και τη δυνατότητα από κοινού να εξετάζουμε θέματα υψής της σημασίας. Και αυτή είναι και η σημερινή περίπτωση της κοινή μας συνεδρίασης θα συζητήσουμε το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πολιετές πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο «Πρόγραμμα της Στοχόλμης» για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Γνωρίζετε ότι όλα ξεκινούν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 10 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για την επόμενη πενταετία, πρώην πρόγραμμα Τάμπερε το 1999 και Χάγη το 2004 στη συνέχεια. 2004 με 2009. Το οποίο λύγει. Και αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης όπως ονομάζεται τώρα αφορά τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ε, στον αστερισμό και τη συνδίκη Λισαβόνας που είναι πιθανότερο από ποτέ να τεθεί σε ισχύ, συνεδριάζουμε σήμερα από κοινού, όπως είπαμε. Τρία μέλη του Κοινοβουλίου επιφορτιστήκαμε με το καθήκον να συντάξουμε ένα ε, κοινό ψήφισμα και να σας υποβάλουμε το σχέδιο. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, στη συνεδρίαση αυτή θα προσκληθούν και μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και προσκαλούνται σε τέτοιες συνεδριάσεις. Γιατί ενισχύεται η συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, στα πλαίσια της Συνθήκης Λισαβόνας. Εξ ονόματος λοιπόν των τριών επίτροπων θα σας παρουσιάσουμε το κοινό ψήφισμα. Κύριε Καζίνη. Ο κύριος Καζίνη είναι εισηγητής ε, της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων. Είναι ο κύριος Μπέλιγκουερ, ε, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και εγώ εξ ονόματος της Επιτροπής Ελευθεριών. Συνεισηγητές οι τρεις. Καταρχάς θα πρέπει να εγκρίνουμε τη μίληση σε διάταξη. Κατάθεση τρόπολογίων μέχρι τις 22 Οκτωβρίου Και τελικά θα πρέπει να εγκρίνουμε και δύο προφορικές ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο για να έχουμε τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Για τη μεταβατική περίοδο. για τη μετάβαση από τη συνθήκη της Νίκαιας που ισχύει αυτή τη στιγμή στη συνθήκη της Λισαβόνας και τη μεταφορά των θεμάτων από τον τρίτο πυλώνα στον πρώτο και όλο το κοινοτικό και εκτιμένο των θεμάτων ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Αν δεν διαφωνεί κανείς λοιπόν με το σχέδιο της τη της διάταξης, θα εγκρίνουμε και προχωρούμε αμέσως στη παρουσίαση της κοινή έκθεσης. Εγώ θα σας παρουσιάσω τα βασικά χαρακτηριστικά. Όπως όλοι γνωρίζετε, η συνθήκη της Λισαβόνας, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ, όσο νούπο, πολλοί από εμά το περιμένουμε εδώ και καιρό αυτό, βάζει τα θεμέλια, τους στόχους και περιγράφει τη μέθοδο εργασίας ε, του λεγόμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Μετά το Ιρλανδικό δημοψήφισμα, η προοπτική αυτή της θέσεως ισχύ της Λισαβόνας έρχεται πιο κοντά μας. Και είναι πιο αξιόπιστη από ποτέ. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα ενίσχυση τη συνεργασία στα πλαίσια του Σέγγεν, όπως έχει αποδειχτεί, βρίσκεται αυτό το κέντρο, στην καρδιά του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το Σέγγεν σημαίνει ακριβώς αυτό, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη στο εσωτερικό ε, της κοινοτικής επικράτειας και εντός των κοινοτικών συνόρων. Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Αλλά όχι μόνο αυτό, σημαίνει και άσυλο, προστασία των προσφύγων, ε, μεταναστευτικές πολιτικές και διαχείριση όλων αυτών και των μεταναστευτικών ρευμάτων και ε, έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ένα δεύτερο σημείο, το οποίο τονίζεται στην έκθεση, που σας παρουσιάζουμε σήμερα το απόγευμα, ε, σχετίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πάρα πολύ σημαντικός πυλώνας είναι αυτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο σύνολό του. Μιλούμε λοιπόν για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι ελευθερίε στην έκθεση, για την προστασία τους τη προστασία τη αξιοπρέπειας και της ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Καλή είναι η καταπολέμηση της ε, ε, εγκληματικότητας, του οργανωμένου εγκλήματος και της αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται και αυτά υπόψη. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι η σημασία Σύνδεση σύνδεσης και συνεργασίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναπτυχθεί πλήρως ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τα επόμενα έτη. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν να τονίσω και αυτό το σημείο, αυτό το σημαίνει ότι εμείς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να λαμβάνουμε ε, πολύ σοβαρά υπόψη περισσότερο από ποτέ τους ίδιους μας τους εαυτούς. Θα πρέπει να πιστέψουμε ότι έχει νέες δυνατότητες, νέες εξουσίες πλέον το Κοινοβούλιο. Είναι συνομοθέτης, συναποφασίζει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να ανακτήσουμε την αξιοπιστία και το σεβασμό μας, να μας σέβονται, να λέμε την άποψή μας, να γίνεται σεβαστή, ε, και η δέσμευσή μας στα μάτια των πολιτών. Πώς θα γίνει αυτό. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι από τα σημαντικότερα ατού αυτά της συνθήκης Λισαβόνας. Συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι μια πολυεπίπεδη δομή εξουσίας αυτή και διαχείρισης και διακυβέρνησης για την εφαρμογή όλων αυτών των νέων νομοθετικών ε, δράσεων. Η καταπολέμηση του εγκλήματος, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το Σέγγεν ως χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Ένα τελευταίο σημείο συνδέεται με την αύξηση της αποτελεσματικότητάς μας, που θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, ε, τα ε, σώματα των νομικών ε, νομομαθών, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι, εκείνοι που εφαρμόζουν και ασχολούνται στην καθημερινή τους επαγγελματική ζωή με τα νομικά, θα πρέπει να συνεργάζονται σε αυτό τον ενισχυμένο χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Είναι όλο και πιο απαιτητική η άσκηση των νομικών επαγγελμάτων παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία αξιολόγησης για καλύτερη εφαρμογή στη συνέχεια των ευρωπαϊκών πολιτικών που αποφασίζουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου τη εφαρμογής όλων αυτών που αποφασίζουμε στον χώρο της ασφάλειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Να ελέγχεται και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα, αλλά και η δικαιοσύνη, το πόσο δίκαιη δηλαδή είναι η δικαιοσύνη στην απονομή τη. Πρόκειται λοιπόν να εγκαταστήσουμε μια νέα δυναμική και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια ετήσια συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. με εστίαση ακριβώς στην εφαρμογή και την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Στον χώρο αυτό των μεγάλο της ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης και στο επίκεντρο πάντα είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Αυτά. Όπως μπορείτε να φανταστείτε και να επαληθεύσετε από τα κείμενα του κοινού σχεδίου ψηφίσματος που σας έχει διανεμηθεί, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και τα κύρια ε, της συνεισφοράς της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Έχουμε ενώπιον μας ένα χρονοδιάγραμμα η προθεσμία για την κατάθεση των απολογιών είναι 22 Οκτωβρίου. Σε άλλη πάλι τέτοια κοινή συνεδρίαση στις 12 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε και έπειτα και άλλη συνεδρίαση όπου επίσημα θα καλέσουμε τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων εδώ στο Κοινοβούλιο στις 16 και 17 Νοεμβρίου. Και τέλος η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στις 23 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν έχει το χρονοδιάγραμμά μας αυτή τη στιγμή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καζίνη για να μας δώσει την άποψη της δικής του Επιτροπής, μετά στον κύριο Μπέλιγκουέρ, στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και θα αρχίσει η συζήτηση. Βέβαια θα πρέπει να ξέρετε ότι στις 4 ώρα πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η διαδικασία, κάπως επιταχυμένη ασυνήθιστα, είναι ασυνήθιστη λόγω της σημασίας του προγράμματος της Στοκχόλμης, που πρέπει να ληφθεί απόψε από το Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου. Γι' αυτό, όπως ε, είπε ο πρόεδρος Αγγιλάρ, απαιτεί εκ μέρους μας αυτή την επιπλέον προσπάθεια. Η Συνταγματική Επιτροπή, τη οποίες προεδρεύω, ασχολείται φυσικά με τα συνταγματικέ πτυχές του προγράμματος. Μέχρι στιγμή κάθε Επιτροπή ετοίμασε ένα σχέδιο κειμένου η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, η Νομική και η Συνταγματική. Τα τρία αυτά κείμενα τα συζήτησαν οι εισηγητές σε μια συνεδρίαση μεταξύ τους κατέληξαν σε ένα ενιαίο κείμενο σε μια δεύτερη συνεδρίαση εκρήφη μακροσκελές είχε 10 σημεία πάνω από 20 σελίδες Γι' αυτό έχουμε το νυν κείμενο που όπως διαπιστώνετε δεν είναι μεν πολύ σύντομο αλλά είναι επαρκώς συνοπτικό. Το τμήμα του εγγράφου αυτού που αφορά την παρέμβαση της Συνταγματικής Επιτροπής θα ήθελα να τονίσω τα εξή. Πρώτον, είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι επεκτείνουν οι νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβουλίου. Με συγκεκριμένο αίτημα προς το Συμβούλιο για τις τρέχουσες διαδικασίες μέσω της διαβούλευσης, ενώ τώρα θα περάσουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα περάσουμε σε ένα κανονικό νομικοθετικό σύστημα, δηλαδή στην απόφαση η διαδικασία να, να ξαναρχίσει από την αρχή με νέα απόφαση στο Κοινοβουλίο. Δεύτερο σημαντικό θεσμικό θέμα που το ανάφερε ο πρόεδρος Αγγιλάρ είναι η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στη δραστηριότητα του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν υποκαθιστά βέβαια ο ρόλος αυτός στην δική μας δραστηριότητα. Είναι ένα εργαλείο περαιτέρω εμβάθυνσης και πιο άμεση συμμετοχή των λαών. Γιατί τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πιο κοντά στους λόγους από ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα μπορούν με την παρουσία τους στην νομοθετική δουλειά και στη λήψη των αποφάσεων του Κοινοβουλίου να παίξουν σημαντικό ρόλο. Έπειτα η αρχή της επικουρικότητας. Πολύ σημαντικό στην εφαρμογή της. Πρέπει με ακρίβεια να ορίσουμε τα όρια τον έλεγχο και τη συμμετοχή των κρατικών ε, των, κυβερνήσεων, των κρατών μελών. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε η συνεργασία να, αυτή να μην επιβαρύνει την ομοθετική διαδικασία. Άλλο σημαντικό θεσμικό σημείο είναι η ενσωμάτωση στη θήκη της Λισαβόνας στις χάρτες των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήδη θυμόσαστε τι αποφασει 13 Δεκεμβρίου του 2007. Ε, λοιπόν, η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σήμερα θα αποτελεί τμήμα της συνθήκης Λισαβόνα. Άρα δεσμεύει όλε τι χώρε. Επίση, στη συνθήκη της Λισαβόνα επιτρέπεται η ένταξη τη Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την προστασία των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου που δεσμεύει όλες τις χώρες, δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ένωσης ήδη έχουν επικυρώσει αυτή τη συνθήκη. Αυτό ενισχύει την νομική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, προστίθεται και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Βέβαια, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα όσον αφορά τι αρμοδιότητε. Και το κείμενο καλεί το Συμβούλιο να μελετήσει το σημείο αυτό για να μην δημιουργηθεί σύγχυση. Επόμενο σημείο. Έτοιμα για συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Eurojust και το Europol για να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος προκειμένου να ενισχυθούν οι εξουσίες αυτών των δύο οργάνων. Επόμενο, καλούμε προς αξιολόγηση και ενδεχομένω η υλοποίηση μια ενιαίου εκλογικού νόμου και ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να προβληματίσει τη δική μας Επιτροπή είναι το θέμα της μετανάστευσης. Το ξέρουμε το θέμα, είναι τεράστιο και χρειάζεται μια προσέγγιση κατά τη γνώμη της Συνταγματικής Επιτροπής όχι μόνο σε βάση συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών, αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ω Ιταλό, ξέρω πόσο απαιτείται αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, ωστόσο θεωρώ ότι απαιτεί μια νέα προσέγγιση θεσμική, γιατί τα σύνορα των κρατών μελών είναι σύνορα τη Ευρώπη. Όποιο μπαίνει στη Σικελία ή στην Ελλάδα ή στην Ισπανία μπαίνει στην Ευρώπη, γιατί η αρχή τη ελεύθερη κυκλοφορία τα επιτρέπει όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ευρωπαϊκό πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε αλλαγή λίγο στην νοοτροπία όσον αφορά το θέμα αυτό. Πριν περάσουμε σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία όσον αφορά είτε την νόμιμη είτε την παράνομη μετανάστευση. Φυσικά με καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και αποδοχή με μέτρο, αλλά γενναιόδορη, αυτών που προσπαθούν να αποφύγουν τη βία, τις διώξεις και το θάνατο. Αυτά ήταν τα σημεία που ενδιαφέρουν τη Συνταγματική Επιτροπή και υπάρχουν στο κείμενο που έχετε πάρει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πρόεδρε Καζίνη. Περνάμε στον πρόεδρο Μπελιγκουέρα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω τη σημασία του ότι για πρώτη φορά συνεδριάζουμε με αυτή τη μορφή σύνθεση. Αυτό δείχνει την σοβαρότητα της πρωτοβουλίας, γιατί το πρόγραμμα της Στοκόλμης, νομίζω, αποτελεί μια σημαντική συνιστόσα των στόχων της οικοδόμησης της Νέας Ευρώπης. Συγχαίρω τις γραμματείες και των τριών επιτροπών που ξόδεψαν αυτές τις ώρε γιατί με τέτοια ταχύτητα κινήθηκαν, προκειμένου να προσφέρουν αυτό το άριστο έργο, έτσι ώστε πολύ σύντομα να έχουμε ένα κείμενο, ένα έγγραφο, που θα το κρίνεται. Ο στόχος μας είναι ισορροπία σε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου μεταξύ της ανάγκης να μιλήσουμε στους πολίτες όχι μόνο με την κρύα γλώσσα του δικαίου, αλλά ορίζοντας έναν ιδανικό στόχο, δηλαδή το να δημιουργηθεί ένας χώρος δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας στην Ευρώπη, που στο κέντρο του να έχει τον πολίτη και να βρεθεί και η ισορροπία μεταξύ αυτού του ιδανικού στόχου και μια σειρά προτάσεων και μέτρων συγκεκριμένων που να ικανοποιούν την ανάγκη, τις ανάγκες μάλλον, στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Πολύ συγκεκριμένα. Γιατί τα ιδανικά πρέπει να τρέφονται με συγκεκριμένη τροφή. Άλλη ισορροπία που αναζητήσαμε ήταν μεταξύ της φυσικής ανάγκης, της νόμιμης ανάγκης για ασφάλεια που σε αυτή την ιστορική στιγμή που ζούμε απαιτούν οι πολίτες από τη δημόσια αρχή να τους δώσει και ταυτόχρονα να αποφύγουμε τον κίνδυνο να γύρουμε πολύ προς μια ανάγκη ασφάλειας που θα έβαζε σε κίνδυνο τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με πολιετούς, πολιετής αγώνες για τους πολίτες, που είναι καταρχήν το δικαίωμα της ελευθερίας. Μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το δικαίωμα στην Ευρώπη της κινητικότητας. Το σημείο Α. Η συνεργασία του Σέγγεν επιβεβαιώνεται ως το κέντρο. Στην αγγλική αυτή διατύπωση όπου σας διάβασα βλέπουμε ποια είναι η βάση της κινητικότητας. Και βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξουν και όλες οι άλλες προϋποθέσεις έτσι ώστε συγκεκριμένα να υλοποιηθεί η κοινωνικότητα. Θα επιστρέψω σε αυτό σε λίγο. Άλλο σημείο που υπογραμμίζεται στην πρόταση ψηφίσματος είναι το ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης δεν είναι μια απλή συνέχεια του προγράμματος της Χάγης τονίζεται ιδιαίτερα ότι το πρόγραμμα της Χάγης ήταν μια θετική επιτάχυνση όσον αφορά την πολιτική κατά του εγκλήματος στη διαδικασία την ποινική και την ανακριτική αλλά επίσης έχει τα στοιχεία από το Συμφωνία του Τάμπερε. Θέλει, θέλουμε Πρέπει λοιπόν να επαναπροσαρμοστούν οι σχέσεις μεταξύ του πολίτη, μεταξύ των πολιτών και μεταξύ πολιτών και της εξουσίας, έτσι ώστε να καλυφθούν όντως οι ανάγκες των πολιτών. Ένα άλλο γενικό θέμα, πριν πω στις λεπτομέρειες, είναι ότι το πρόγραμμα της Χάγης ότι έχουν γραφτεί πολλά πράγματα τα οποία όμω στην πράξη δεν έχουν υλοποιηθεί. Ωστόσο, στην Ευρώπη, συχνά και στις χώρες μέλη, στις... έχουμε τις διάφορες διατυπώσεις, αλλά δεν έχουμε την πράξη μετά. Και έτσι μειώνεται η αξιοπιστία, η δημοκρατική αξιοπιστία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών που θέλουν να βλέπουν facts, γεγονότα. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό δεν αρκεί να προβλέπουμε νομοθετήματα και μανιφέστα πρέπει να είναι κάτι που να μπορεί να εφαρμόζεται και πρέπει να κάνουμε και μία αξιολόγηση, μία παρακολούθηση του τι συμβαίνει. Και αυτό ζητάμε. Σας διαβάζω στα αγγλικά περιοδική αξιολόγηση των, του ό,τι έχει επιτευχθεί. Πρέπει δηλαδή αυτά να ελέγχονται. Να δούμε έγιναν ή όχι και αν υπάρξουν αποτυχίες, με είναι φυσιολογικό και αυτό, να διορθωθεί η γραμμή πλεύσης. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Το πρώτο σημείο που υπάρχει στη συνθήκη του Στρασβουργού για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα στην αστική δικαιοσύνη που σημαίνει απλούστευση. Περί αυτού μιλάμε. Ο πολίτης χάνεται μέσα στους μεάνδρους, τους νομικούς και τους διαδικαστικούς και στους μηχανισμούς της δικαιοσύνης. Καλύτερη πρόσβαση λοιπόν και να δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα. Είσαι αφορά την επιχείρηση, είσαι αφορά την εργασία, είσαι αφορά την ζωή του πολίτη, είσαι αφορά την αστική, ας το πούμε, τα αστικά θέματα, ή την οικογενειακή ζωή. Το θέμα ε, του διαζυγίου, χωρισμός, οικογενειακό δίκαιο, οι συνθήκε κατά τις οποίες ζουν τα παιδιά, Όλα αυτά αποτελούν βάση της ενιαίας Ευρώπης. Και έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ζουν αυτά σήμερα και δεν πρέπει να θεωρούνται τα σύνορα ενός κράτους κάτι το οποίο να απαγορεύει την κινητικότητα. Έπειτα, για τους καταναλωτές. Και αυτούς τους αφορά η Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. οικονομικά θέματα, εμπορικά θέματα. Ε, το πιστοτικό σύστημα των τραπεζών, το θέμα του company law, του εταιρικού δικαίου, γιατί υπάρχουν κενά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα έχει επισημάνει. Γι' αυτό που αφορά πιο άμεσα θέματα αστικού δικαίου, πρέπει να καλυφθούν και εδώ τα κενά που ήταν στη Ρώμη 2, ο κανονισμός για τη Ρώμη 2. Όπως βλέπετε όλα αυτά είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένα γιατί ο χώρος της δικαιοσύνης συναπαρτίζεται από το όλα αυτά τα σημεία και τη σωστή λειτουργία τους. Έπειτα, εναρμόνιση προκειμένου να είναι συμβατοί οι κανόνες πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Το δικαίωμα όσον αφορά τις διάφορες συμβάσεις και συμφωνίες. Να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα να μην μπλοκάρονται από μια νομοθεσία που είναι διαφορετική και να χρειάζεται να κάνουν σάλτο μορτάλε από χώρα σε χώρα προκειμένου να ακολουθήσουν την νόμιμη λειτουργία τους. Ένα ευρωπαϊκό δίκαιο λοιπόν. Αναφέρονται διάφορες δυνατότητε για κωδικοποίηση, η επιλογή τη εθνικής διαδικασίας, αλλά αυτά θα γίνουν βαθμιαία, βαθμιαία, προοδευτικά και βαθμιαία, όχι εντελώ απότομα. Άλλο θέμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια δικαιοσύνη ευρωπαϊκή εντός εισαγωγικών μονολυθική. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αντίστοιχη κουλτούρα και ενωτροπία Έχουμε δικαστές, δικηγόρους, νομικούς που ίσως και να μην γνωρίζουν πολλά θέματα που συζητιώνται και επιλύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δικαστές και δικηγόρους που γνωρίζουν μόνο τη χώρα τους και δεν ξέρουν τι γίνεται στις άλλες χώρες μέλη. Αυτή η έλλειψη γνώσης, γιατί έχουμε ε, διδαχή της νομολογίας στα πανεπιστήμια, αλλά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο είναι ένα πολύ μικρό, κομματάκι μόνο της διδακτέας ύλη. Και δεν Τη στιγμή όμως παράλληλα αυτή έχουμε παράγγελες κινήσεις μεταξύ του εθνικού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου και αγγελεπίδραση. Πρέπει λοιπόν ακόμα και όταν κάποιο λειτουργεί σε εθνικό κράτος, να γνωρίζει τι γίνεται στην Ευρώπη. Χρειάζεται όμως μια ενεργητική πολιτική σε αυτή της κουλτούρας. Έχουν γίνει μερικά πράγματα, η κίνηση όμως είναι πάρα πολύ αργή. Η Κομισιόν και το Συμβούλιο, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να παρεύουν με συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουν αυτή την ανταλλαγή. Και όπως είπε ο μεγάλος ομονιστής ο Έρασμος, όταν μιλούσε για την Ευρώπη όπου οι εργαζόμενοι θα κυκλοφορούν, ε, αυτό τώρα περνάει και στη σφαίρα του δικαίου. Γνώση των διαφόρων νομικών συστημάτων και η εμπιστοσύνη που έχει μία χώρα για το νομικό σύστημα της άλλης. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, οι αποφάσεις θα είναι σωστές. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, ό,τι και να επιβάλλουμε από πάνω, δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή των ανθρώπων. Αυτή την εμπιστοσύνη λοιπόν πρέπει να προωθήσουμε με τέτοιου είδους μέτρα. Μπορούμε λοιπόν να υποβάλλουμε ένα πρόγραμμα Στοκχόλμης για τον κοινό αυτό χώρο, δικαιοσύνη, ασφάλεια, ελευθερία, που θα είναι βέβαια και ο μεγάλος στόχος για την Ευρώπη, το ιδανικό, αλλά και θα έχει την ικανότητα ο πολίτης να το νιώσει μέσω των πλεονεκτημάτων που θα έχει από την ύπαρξη αυτού του κοινού χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα γίνουν γρήγορες αντιδράσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουμε ε, ήδη έναν κατάλογο 15 και παραπάνω ευρωβουλευτών που έχουν ζητήσει το λόγο οπότε θα πρέπει να σεβαστούμε ε, το χρονοδιάγραμμά μας και γι' αυτό σας εκλυπαρώ να μην ε, ξεπεράσετε τα τρία λεπτά ο καθένας. Εν ονόματι του Συμβουλίου ο κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε τρία λεπτά βέβαια Μπορώ καταρχήν να χαιρετήσω τις τρεις επιτροπές και να τους πω πόσο χαίρομαι και πόσο αισθάνομαι ότι με τιμάτε να συμμετέχω σε αυτή την ε, πρώτη ε, συνεδρίαση μίας μακριάς διαδικασίας που ε, θα ενισχύσει τις επαφές που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δύο υπουργοί μου σας, υπενθυμίζω ήταν στο Κόσαξ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ο Υπουργός μου θα έρθει τον Νοέμβριο και πάλι εις ε, την Επιτροπή σας ε, το Νοέμβριο. Ε, πάντοτε θεωρούμε και επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της Στοκχόλμης το οποίο θα κοιτάζει προς τα εμπρός και θα είναι ισοσκελισμένο. Νομίζω ότι ο κύριος Μπερλίνγκουερ πολύ σωστά εξέφρασε τι ε, επιζητούμε με αυτή την ισορροπία. Θέλουμε ίσως να ε, εξισορροπήσουμε λιγάκι την ε, συζήτηση ασφαλείας και να κοιτάξουμε τα θέματα της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και συγχρόνως να αποφύγουμε μία απειλή ασφαλείας στην Ευρώπη. Όσον αφορά την συνθήκη της Λισαβόνας όπως ελέγχθη στην Επιτροπή Ελευθεριών ότι προημερών δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας ακόμη αλλά όταν θα έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία της Στοκχόλμης θα είμαστε πιο ασφαλείς του θέματος. Ε, θα Πρέπει λοιπόν ε, ε, ακόμη να, γράψουμε το πρόγραμμα διότι έχουμε ξεκινήσει τις ε, διαβουλεύσεις. Έχουμε ακόμη να κάνουμε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Αλλά από ανάγκη και από πεποίθηση θεωρούμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε τα βασικά δικαιώματα, την ε, προσχώρηση προς ε, την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, να τονίσουμε τα δικαιώματα των ατόμων, να υπάρχει αξιολόγηση, όχι τόσο παρακολούθηση, όσο αξιολόγηση, δηλαδή ανταλλαγή των βελτίστων πρακτικών και ε, αμοιβαία ενημέρωση και εφαρμογή. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε την ε, διαφάνεια, το, την ειλικρίνεια, πράγμα το οποίο επιζητούμε και στην νομοθετική διαδικασία και σε άλλα σημεία. Για αυτό το χρόνο λοιπόν απλώς ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι που είμαι εδώ, θα ακούσω πολύ προσεκτικά όλες τις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Νίλσον, ο κύριος Ντεμπράουερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Χάνς είπε ορισμένα πράγματα τα οποία εκπροσωπούν από κοινού και την Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στο γεγονός της ε, γνωμοδότησης που θέλει να εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συμμετοχή του Κοινοβουλίου ή στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Όπως ξέρετε, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Ιουνίου στην παρουσίασή της είχε εμπνευστεί από αυτές τις ιδέες και αυτές οι ιδέες βρίσκονται στο προσχέδιο του ψηφίσματος που θα αποτελέσουν τη βάση των, συζητήσεών σας εφ' εξής βασιζόμαστε στο πρόγραμμα της Χάγης, όχι όμως μόνο σε αυτό. Ε, βασιζόμαστε συγχρόνως σε ένα σαφές όραμα των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επομένη πενταετία, είτε πρόκειται για τους πολίτες, είτε πρόκειται για τις εξελίξεις ενός κοινού χώρου δικαιοσύνης, ανοίγματος προς μία νέα προσέγγιση της, πραγματο... της πραγματικότητας, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις ροές των μεταναστών. Όταν θα ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας θα υλοποιηθούν όλα αυτά, αλλά ελπίζουμε ότι θα μπορέσει σύντομα να εφαρμοστεί η συνθήκη ε, και οι πολιτικές αυτές θα συμβάλλουν στο να επιταχυνθεί η υλοποίηση της συνθήκης Λισαβόνας. Γι' αυτό ε, για τις συνθήκη του Άμστερνταμ θεωρήσαμε ότι αυτή συνέβαλε εις την πρόθεση των θεμάτων που πραγματευόταν ε, θέλουμε να υπάρχει περισσότερο δημοκρατικός έλεγχος, ενισχυμένος έλεγχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτό θα ε, συστεί ε, σε κοινέ μας δράσεις. Γι' αυτό ο πολίτης θα αποτελέσει το επίκεντρο των μέλημάτων μας. Αυτός είναι, αυτή είναι και η επικεφαλίδα της ανακοίνωσής μας. Θα πρέπει να ε, εντοπίσουμε τις πραγματικότητες που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προβλήματα που έχει να επιλύσει, θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία και να υπάρχει συνεργασία πιο ενισχυμένη. Πρέπει να πω ότι η πρώτη ανάγνωση του προσχεδίου στο οποίο θα βασιστούν οι εργασίες μας μας οδηγεί στο να θεωρήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν κοινά μελήματα. Ωραία, τώρα θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τους ε, ευρωβουλευτές αλλά ζήτησαν και άλλοι δύο ευρωβουλευτές το λόγο. Είχαμε πει ότι είχαμε ήδη 15 και έτσι τώρα κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών και το λόγο έχει ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως διότι μας συγκεντρώσατε όλους μία πέμπτη απόγευμα με τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων και χαιρόμαστε για τη συνεργασία. Εν ονόματι του ΕΛΚ κύριε ε, Πρόεδρε πρέπει να σας πω ότι το ΕΛΚ προσβέπει σε μία Ευρώπη των πολιτών πιο ασφαλή και αμέσως τονίζω την ασφαλή Ευρώπη γιατί βλέπω από το προσχέδιο του ψηφίσματος ότι ε, το κείμενο έχει ε, κάπως ε, αποδυναμωθεί. Αυτό το σχέδιο πήραμε τώρα, δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς, αλλά θεωρούμε ότι η Ευρώπη των πολιτών πρέπει να είναι και ασφαλέστερη και γι' αυτό το ΕΛΚ στηρίζει το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Θέλουμε ρεαλιστικό και συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα σαφή χάρτη πορείας για την επόμενη πενταετία για να καταρτήσουμε ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας και να επικεντρώνεται στους πολίτες. Όχι μόνο δηλαδή να δημιουργηθεί ο χώρος, αλλά ε, να προσφέρουμε αυτό το χώρο στους ε, πολίτες που χρειάζονται περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη ασφάλεια. Χρειαζόμαστε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Χαιρετίζουμε λοιπόν εμείς τουλάχιστον το αποτέλεσμα της Ιρλανδίας, ιδίως στα θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης, θα μπορέσουμε ε, να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συναδέλφους στα Εθνικά Κοινοβούλια και χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων και γι' αυτό είναι καλό διότι η συνθήκη αυτή για πρώτη φορά ε, διατυπώνει τις αρχές αυτές συγκεκριμένα. Θα πρέπει όμως επίσης να συγκεκριμενοποιήσουμε δύο θέματα. Πρώτον την αλληλεγγύη και δεύτερον την επικουρικότητα. Όσον αφορά την αλληλεγγύη στο τομέα μετανάστευσης και ασύλου απέχουμε ακόμη πάρα πολύ από το να επιτύχουμε συγκεκριμένη αλληλεγγύη ακόμη και μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πόσο μάλλον με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει αλληλεγγύη, πραγματική, ενεργή και όχι μόνο στα λόγια. Χρειαζόμαστε και επικουρικότατα. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να εμπλεκόμαστε όταν ε, έχουμε αρμοδιότητα. Αλλά δεν θα πρέπει ε, να εμπλεκόμαστε εάν δεν υπάρχει αρμοδιότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει στο εθνικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν μια τεράστια πρόκληση, πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω ότι όλοι θα εμπλακούμε σε αυτή τη διαδικασία και θα θελήσουμε να συμμετάσχουμε για να μπορέσουμε πραγματικά να επιτύχουμε έναν χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης ε, και ασφαλείας. Ο κύριος Μωράης για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με το πνεύμα το οποίο έκανε γενικές παρατηρήσεις ο κύριος Μπουσουτήρη θα κάνω και εγώ διότι ε, αυτές ε, οι, ε, αυτό το ψήφισμα είναι ένα πολύ ισοσκελισμένο κείμενο, διότι όπως είπε και ο κύριος Μπουσουτήλ, πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι μας είπε ο κύριος Λοπές ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 είναι μια ιδιάζουσα συνεδρίαση και αυτό το οποίο θα γίνει τώρα με, τις εθνικές, με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τις συνθήκες της Ξαβώνας είναι πιο σημαντικά Άρα ο χάρτης πορείας που ανέφερε ο κύριος Μπουσουτήλ παίρνει μεγαλύτερη σημασία. Θα πρέπει να είναι ποιοτική κάθε παράγραφός του. Αν αναφερθώ στην αλληλεγγύη, το άσυλο και τη μετανάστευση, αν δείτε τις παραγράφους της μετανάστευσης υπάρχει μία ισορροπία, αλλά υπάρχουν και σημεία κλειδιά τα οποία θέλουν τροποποίηση, διότι μιλάμε για την αποφυγή των νέων συστημάτων όπου υπάρχουν ήδη συστήματα και προστασία δεδομένων. Χρειαζόμαστε όμως και νέα θέματα από πλευράς αλλήλου. Ήθελα λοιπόν αυτό το παράδειγμα να μπορέσει να σκιαγραφίσει ότι στο κείμενο αυτό πολλά πράγματα χρειάζονται αλλαγή αλλά ουσιαστικά είναι ένα ισορροπημένο κείμενο σωστός χάρτης πορείας που ε, ε, ε, διατυπώνει Λοιπόν, τα δικαιώματα του ατόμου και τα δικαιώματα όσων θέλουν να έρθουν στην Ήπειρο αυτή. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο να διατηρήσουμε τις ισορροπίες μετά την Λισαβόνα. Ελπίζω λοιπόν ότι η πολιτική μου ομάδα, η σοσιαλιστική, θα μπορέσει να διατυπώσει τροπολογίες στις λεπτομέρειες ε, ε, μέχρι τέλος Οκτωβρίου και ελπίζουμε το κείμενο αυτό θα ισχύσει για πέντε χρόνια και θα είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Για τρία λεπτά. Πρόεδροι, σας ευχαριστώ που διοργανώνετε τη συνεδρίαση αυτή. Είναι αρκετά ενδιαφέρον πείραμα, θα έλεγα, συνεργασία τριών επιτροπών που έχουν διακριτή φιλοσοφία και ε, κουλτούρα και ευθύνη η καθεμιά. Ε, πάντως, νομίζω θα είναι ένα πρώτο πείραμα στο καθήκον που έχουμε, το θεσμικό, να συνεισφέρουμε στον κοινό προγραμματισμό. Κοινό και εδώ εννοώ μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, ε, Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το πώς ε, χαράζουμε την ημερησία διάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να εκλειφθεί και ως προπαρασκευαστική συνεδρίαση για τις ακροάσεις των επιτρόπων που είναι αρμόδιοι για ε, τον χώρο αυτό ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και θα αναλάβουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια και οι ακροάσεις θα γίνουν το Δεκέμβριο. Αν είμαστε τότε σε θέση να διορίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να φέρω μερικά σημεία αναφερόμενος στη συνταγματική πτυχή του κοινού ψηφίσματος. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία μιας διαδικασίας ε, πώς να το χαρακτηρίσω ε, όπου να μπορεί κανείς να τραβάει φρένο επιγόντως δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τροχοπέδες δεν υπάρχουν ε, ε, δυνατότητες διακοπής κάποιες διαδικασίες. Αλλά αν εφαρμοστεί η διαδικασία αυτή, οι πρωτοπόροι και ενδιαφερόμενοι περισσότερο θα ε, έχουν ε, μια φυγή προς τα εμπρός και θα έχουν ένα είδος ενισχυμένης συνεργασία. Και είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προετοιμάσουμε και το Συμβούλιο να αντιμετωπίσουμε την περιπλοκότητα της πρόοδου ε, κάποιων πυρήνων ε, κάποιων κρατών που είναι ε, και πιο γρήγορα αλλά και ε, έχουν και πιο φεντεραλιστική νοοτροπία και τάση. Αυτό ήταν το ένα θεσμικό, το συνταγματικό. Το δεύτερο, τι γίνεται με τα opting out τις εξαιρέσεις. Από εκεί έρχεται να προσθεθεί αν είναι σωστή αυτή η ορολογία, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδική Δημοκρατία. Όλη αυτή η ιστορία για την εσωτερική δικαιοσύνη και τη στρατηγική καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει κατά την άποψή μου να συνδέεται περισσότερο και πιο άμεσα με την στρατηγική εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λείπει αυτή τη στιγμή από το κοινό ψήφισμα και είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να δούμε στο μέλλον αυτό. Θα ήθελα επίσης να επιμείνουμε περισσότερο και σε μεγαλύτερο βάθος στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των αποφάσεων του ε, ΔΕΚ, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Θα τα δούμε αυτά στο μέλλον. και κατά πόσο αυτό θα έχει κάποια μαγική συνέπεια στην ποιότητα των πολιτικών και στην ανταπόκριση των πολιτών στις πολιτικές αυτές. Ίσως επίσης να βοηθούσε εάν ε, τονίζαμε και πάλι ρητά τα καθήκοντα εδώ και τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων. Νομίζω εξηγήθηκε αυτό το θέμα από τον πρόεδρο κάπως γενικά και αόριστα. Ως εισηγητής για τη μεταρρύθμιση ε, ε, του εκλογικού συστήματος στο Κοινοβούλιο, θα πρότεινα να προσθεθεί και άλλη μια παράγραφος, η οποία να προβλέπει τις οποίες μεταρρυθμίσεις θα έχουμε ε, και προβλέπουμε στη Συνταγματική Επιτροπή. Και τέλος, με μεγάλο σεβασμό προς την Προεδρία, πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μένουμε ικανοποιημένοι με την απλή ιδέα της αξιολόγησης και μόνο του συστήματος. Ο χώρος ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης μεγαλώνει, διευρύνεται και ειλικρινά πιστεύω ότι ο έλεγχος, η παρακολούθηση, το monitoring αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι απλή αξιολόγηση. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό ενός συστήματος, όπου, από ό,τι φαίνεται, ορισμένοι πρωθυπουργοί θεωρούν ότι ήδη ε, είναι ε, πρώτη, ε, όχι ίση μεταξύ όλων, αλλά πρώτη μεταξύ όλων. Πρίμου σούπερ πάρεις και όχι πρίμου σύντα πάρεις. Η κυρία Γόλης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συγγητές Εγώ είμαι εκ μέρους της Επιτροπής Αναφορών εδώ. Που κανονικά θα πρέπει να είναι συντάκτη γνωμοδότηση. Εξ τη Επιτροπή μα, λοιπόν, και επειδή είμαι φυσικά και μέλο τη Νομική Επιτροπή, θα σα μιλήσω. Εκ μέρου καταρχήν τη Επιτροπή Αναφορών, υποβάλαμε ένα έγγραφο εργασία που στηρίζεται σε πολλές αναφορές και αιτήσει πολλών ετών θέμα θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας και επισημαίνει τους τομείς όπου οι πολίτες θεωρούν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και που χρειάζεται παρακολούθηση και δεν υπάρχει επαρκής σωστή εφαρμογή. Η Επιτροπή Αναφορών λοιπόν θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε στεναροί, σκληροί στο θέμα αυτό. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές και εγώ επικροτώ την ισορροπία που επετεύχθη με το έγγραφο αυτό. Δέκα χρόνια έχω ευρωβουλευτή και πρώτη φορά βλέπω ένα κείμενο για το θέμα αυτό, ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία, που σωστά δίνει το χώρο που χρειάζεται για την ε, αστική δικαιοσύνη και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Μπελιγκοέρ, διότι όντω θέλουμε να έχουμε στο κέντρο του ενδιαφέροντό μα τον πολίτη. Αν θέλουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που να είναι απλό, διαφανές και κατανοητό για τον πολίτη, πρέπει κάτι να πούμε και για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα προβλήματα των opt-out, δηλαδή εγώ δεν παίρνω μέρος σε αυτό και διάφορα άλλου είδους τέτοιες ρυθμίσεις. Διότι υπάρχουν προβλήματα. Μέχρι στιγμή το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα απλώ να πει ναι σε θέματα διεθνούς δικαίου, σε θέματα που αποφασίζονται στη διάσκεψη της Χάγης. Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με εθνικά κοινοβούλια να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή και γι' αυτό ελπίζω αυτό να μπει κάπου μέσα στο κείμενο. Δικαιώματα των πολιτών. Μία παράγραφος λέει μιλάει για τα δικαιώματα των παιδιών. Νομίζω ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει την εμπειρία του Κοινοβουλίου πρέπει να πούμε κάτι εντελώς χωριστά, σχεδόν χωριστή παράγραφος για τα δικαιώματα του παιδιού και εμπειρίες ε, ζευγών, ε, είτε παντρεμένων είτε όχι, που χωρίζουν και τι συνεπάγεται αυτό. Άσκηση των δικαιωμάτων της ε, υπηκότητας. Δίνουμε δυνατότητα στα δημοκρατικά δικαιώματα των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ας δώσουμε και χώρο και στον πολίτη να πούμε κάτι παραπάνω για τις αναφορές, αλλά το πιο σημαντικό, τώρα που είμαστε στο σωστό δρόμο, είναι να πούμε κάτι για την πρωτοβουλία των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Κάτι πρέπει να πούμε γι' αυτό, για την ευρωπαϊκή υπηκότητα. Από την εμπειρία της Επιτροπής μας πάλι, αυτό που λέει το προτινόμενο ψήφισμα για την ελευθερία κίνησης των πολιτών είναι αρπαρκές. Μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Επίσης, πρέπει κάτι παραπάνω να πούμε για το θέμα της νομικής και δικαστικής εκπαίδευσης. Βέβαια είναι θέμα κρατών μελών, αλλά διστάζουν οι χώρες μέλη να εκπαιδεύσουν στο ευρωπαϊκά δικαστικά θέματα. Πρόεδρος, η Γερμανική Βουλή έχει, θα έχει τώρα το λόγο, αλλά σας θυμίζω ότι μάξιμουμ τρία λεφτά σας παρακαλώ. Ο κάθε μιλητής, η κυρία Ντίκμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω διότι και οι εθνικοί βουλευτές έχουν εδώ τη δυνατότητα σήμερα να παρέμβουν και ουσιαστικά ήδη προκαταλαμβάνουμε τη Λισαβόνα και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό. Χαίρομαι επίσης διότι η Ιρλανδία έχει υπερψηφίσει το δημοψήφισμα για τη συνθήκη της Λισαβάνας και ελπίζω ότι γρήγορα θα υπάρξουν οι τελευταίες κυρώσεις για να μπορέσουμε να έχουμε πιο συχνά να μία τέτοια ανταλλαγή μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε αυτό να το επαναλαμβάνουμε πιο συχνά. Και αυτό θα κάνει πολύ καλό στην ε, αποδοχή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Είμαι εκπρόσωπος των ε, φιλελευθέρων της Γερμανίας και θα αναφερθώ η νομική η πτυχή της ε, ε, δικαιοσύνης. Δηλαδή στο μέλλον ο κύριος Μπαρόζο ε, θα έχει δύο επιτρόπους, έναν για τα εσωτερικά και έναν για τη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι αυτό θα είναι πολύ καλό για τους τομείς αυτούς. Χαίρομαι που θα συνεχιστεί η συνεργασία αλλά η επικουρικότητα και η αναλογικότητα ελπίζω θα λάβουν την προσοχή που τους αποδίδει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θίγησαν και θα πρέπει καταρχήν να, λειτουργήσουν και στα κράτη-μέλη, να εφαρμοστούν. Γι' αυτό και σας παρακαλώ να λάβουμε υπόψη και το γεγονός αυτό. Δηλαδή να μην ε, υπάρξει μία σειρά φακέλων οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο και δεν έχουμε αποκομίσει κάποια πείρα να αλλάξουν. Ε, να τροποποιηθούν. Για μένα είναι πολύ βασικό ότι θα έχουμε ε, πάρα πολλά ε, κατώτατα όρια σχετικά με τα δικαιώματα των εναγωμένων διότι χωρίς αυτά δεν θα μπορέσει να υπάρξει αρμόνιση και αμοιβαία αναγνώριση. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα για τους εναγωμένους διότι εδώ και 10 χρόνια το θέμα αυτό υπάρχει στην ε, ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν έχουμε προχωρήσει και ελπίζω ότι το πρόγραμμα της Στοχόλμης θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή του συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο όσον αφορά την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ε, εμπράγματο δίκαιο νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά διότι η συνθήκη της Λισαβόνας είχε σαφές επιταγές τις οποίες δεν πρέπει να υπερβούμε. Το ποινικό δίκαιο δεν πρέπει να είναι παρά μόνο η τελευταία προσφυγή και θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν ε, υπάρχουν ε, μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την μορφή και το μέτρο της ποινή ε, να προσέξει κανείς πάρα πολύ σε τι θα χρησιμοποιήσει για την ε, ε, νομοθεσία πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να διασφαλίσουμε την αμοιβαιότητα της εφαρμογής διότι διάβασα στο υπόμνημα ότι ζητείται ένα ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά το, ε, ε, το ε, εταιρικό δίκαιο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ούτε προβλέπει μια τέτοια αρμοδιότητα για την Ευρώπη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ διότι το πλαίσιο αναφοράς μας δίνει καλή δυνατότητα να καταστήσουμε πιο ενιαίο το δίκαιο διότι το δίκαιο πολλές φορές η δικαιοσύνη είναι κάτι το δυσνόητο για τους πολίτες και θα πρέπει να ανακοινώσουμε ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω επιμόρφωση των ε, δικαστών και ολόκληρου του προσωπικού της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ, αλλά τρία λεφτά παρακαλώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, και τους ε, τρεις συζήτητες που από ό,τι φαίνεται προσπάθησαν στις εργασίες τους να ανταποκριθούν και στα όσα λένε οι επιτροπές τους. Στην κοινή πρόταση υπάρχουν και κάποια θετικά. Η παραπομπή, ας πούμε, στο πρόγραμμα του Τάμπερε. Η, ε, η ρίση ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό το πνεύμα. Να είναι στο επίκεντρο πάντα τα δικαιώματα των πολιτών. Και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να πω το εξή, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία που ε, πολλοί την ανέφεραν και πάντα αναφέρεται, μια ισορροπία ανάμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα και στα συμφέροντα ασφαλείας. Νομίζω ότι εμείς ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβληματιστούμε. Υπάρχουν θεμελιώδη δικαιώματα που είναι απόλυτα όμως και αδιαπραγμάτευτα και κάθε ισορροπία έχει και τα όρια τη. Δεν θα πρέπει όλα να υπόκεινται και να ζυγίζονται με βάση την ισορροπία. Είναι σωστό να βάζουμε στο κέντρο το πολίτη, αλλά είναι λάθο να το βάζουμε μόνο στο κέντρο τη ασφάλεια. Και όχι στο κέντρο των ιδίων του προσωπικών δικαιωμάτων, ατομικών δικαιωμάτων. Νομίζω εδώ υπάρχει ανισορροπία. Ακριβώ διαταράσσεται η ισορροπία. Διότι όλο και περισσότερο έχουμε γενικά μέτρα προληπτικά εγκάρσια έναντι όλων και απέχουν και περισσότερο από μεμονωμένες δικαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στην πολιτική ασφαλείας. Όλα αυτά συνδέονται με απλές υποψίες. Δηλαδή, τελικά δεν θα πρέπει να ε, είναι ε, ανάλογοι ε, η εφαρμογή των μέτρων που σωστά λέει η έκθεση, αλλά και τα ίδια τα μέτρα που συζητάμε, τα ίδια τα νομοθετήματα, θα πρέπει να ε, ε, έχουν κάποια αναλογικότητα και σε αφηρημένη μορφή, όχι μόνο στην εφαρμοσμένη. Και έχουμε την εντύπωση ότι δεν διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η ισορροπία της ασφάλειας αφενός με τα δικαιώματα των πολιτών, ανδρών και γυναικών αφετέρου. Και στην κοινή σα έκθεση, α πούμε, βλέπω τι γίνεται με την προστασία των δεδομένων, την προστασία τη ιδιωτική ζωή δεν έχουν όλα αυτά τη θέση που τους αρμόζει. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις βάσεις δεδομένων των συστημάτων προφόρησης που έχουμε στην Ευρώπη, που ε, όσο ε, περνάει ο καιρός αλληλοσυνδέονται, αλληλοδικτυώνονται. Μα υπάρχουν κάποιες βάσεις δεδομένων που ε, καταρτίζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει στο μέλλον να έχουν πρόσβαση ε, οργανισμοί ασφαλείας τύπου Ευρωπόλ κατά το δοκούν στη Γερμανία. Έχουμε ε, με τα λόγου γνώσεως διαχωρίσει τις μυστικές υπηρεσίες από την αστυνομία και καλό θα είναι αυτό να γίνει και παντού στην Ευρώπη και να το συζητάμε και συγκεκριμένα πώς θα γίνει. Επιτέλους, ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να βάλουμε και όρια στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας να μην ε, ε, οδηγούμαστε προς μια γενική υποψία, να υποπτευόμαστε όλους τους πολίτες. Δεν οφείλει ο πολίτης να αποδεικνύει την αθωότητά του, αλλά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ε, το κράτος και οι κρατικές δομές θα πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι απαραίτητα. Και εγώ δεν βλέπω ούτε συγκεκριμένες αποδείξεις, ούτε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα μέτρα αυτά εφόσον δεν μας το έχετε αποδείξει αυτό. Ο κύριος Μποργέτσιο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μερικά σύντομα σχόλια. Στο βαθμό βέβαια που δυστυχώς για μια φορά ακόμα στην Επιτροπή Ελευθερών τα έγγραφα έρχονται την τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνω τις, τους λόγους και τις δικαιολογίες, αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική συνεδρίαση, το ότι το έγγραφο το πήραμε την τελευταία στιγμή και όχι μεταφρασμένο είναι πολύ σοβαρό. Δεν δικαιολογείται. Τα σχόλια μου τώρα. Δεν μας αρέσει το ότι στο, στο κείμενο της Στοχόλμης δεν τονίζεται ιδιαίτερα με τα μεγάλα θέματα όταν μιλάμε για ασφάλεια, τρομοκρατία και πιο συγκεκριμένα τον τρομοκρατία που σχετίζεται με τον Ισλαμικό φονταμεταλισμό και να προσαρμοστεί η νομική και δικαστική απάντηση που πρέπει να δοθεί στο περίπλοκο αυτό φαινόμενο και στην ε, τρομοκρατική απειλή που προσαρμόζεται, προσαρμόζεται συνεχώς και τεχνολογικά. Η διείσδυση στις ε, οργανώσεις των τρομοκρατών θα έπρεπε να επιστήσει πολύ περισσότερο την προσ... πολύ περισσότερο την προσοχή μας. Όπως επίσης και η σχέση μεταξύ τρομοκρατικών και εγκληματικών οργανώσεων και λαθρεμπόριο μεταναστών. Είναι θέμα ευαίσθητο, είναι θέμα ταμπού. Πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά, σαν χειρούργοι. Δεύτερο, αποδίδω τιμή στον πρόεδρο Μπελγινγκουέρ στο ότι υπογράμμισε ιδιαίτερα τα πράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα έλεγα περισσότερο τα δικαιώματα αυτών που δεν έχουν τα χρήματα για να προσφύγουν στην αστική δικαιοσύνη. Πολύ σημαντικό. Στην Ιταλία και σε άλλε χώρε, φαντάζομαι, στοιχίζει πάρα πολύ να χρησιμοποιήσει κανεί την αστική δικαιοσύνη και εκατομμύρια πολιτών και καταναλωτών και χρηστών μένουν μακριά υφίστανται λύσεις σε βάρος τους γιατί δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε ένα τέτοιο μακρό πρόγραμμα ζωής που να μπορούν να ε, αντέξουν μέχρι πέρας μια δικαστική διαδικασία που παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Η Ευρώπη στα λόγια προσπίζει τις μειονότητες. Όταν όμως πάμε να εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα βλέπουμε τη δυσκολία. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει στο δικαστήριο στη γλώσσα του. Μια εθνική μειονότητα, γλωσσική. Και ουσιαστικά σιγά σιγά πνίγουμε την νομική ταυτότητα των πολιτών μας. Υπάρχει ένα παραδοσιακό δικαίωμα, παράδοση, δικαίωμα των πολιτών και το ευρωπαϊκό υπερκράτος πάει να το σκοτώσει, να το πνίξει. Έχουμε την υποχρέωση να το προσπίσουμε αυτό με νύχια και με δόντια. Ο πρόεδρος ζητάει τον μιλητή να σταματήσει. Ε, δεν αναφέρονται τα δικαιώματα των θυμάτων, άλλο ένα κενό στο κείμενο. Δεν αναφέρονται τα δικαιώματα αυτά. Δεν μιλάμε για τα δικαιώματα του Άβελ, μιλάμε για τα δικαιώματα του Κάιν μόνο. Η κυρία Φλότρα, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για αυτή την κοινή πρωτοβουλία που μας επέτρεψε να κάνουμε αυτή εδώ τη συζήτηση για μια σημαντική πρόταση της Κομισιόν με ετήσιο πρόγραμμα και πολλές νομοθετικές προτάσεις. Αυτός ο χώρος ελευθερίας ασφάλειας δικαιοσύνης έχει σαν στόχο τα θεμελιώδη δικαιώματα να τα ζουν και να τα απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Και δεν εννοώ μόνο τους πολίτες με τη στενή έννοια του όρου. Όλα τα πρόσωπα, όλοι οι άνθρωποι. Οι πολίτες όπως τους ορίζει η Λισαβόνα είναι πολίτες της Ένωση, είναι πολίτες μιας χώρας μέλος. Αυτό είναι πολύ περιοριστικό ως ορισμός. Υπάρχουν οι άνθρωποι όλοι που ζουν στην επικράτεια της Ένωσης και πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διατύπωσή μας αυτή. Παραδείγματο χάρη, στην παράγραφο που αναφέρεται για την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης που κατά τη γνώμη μου τα αντιμετωπίζει μεροληπτικά η Κομισιόν. Γιατί από τη μια μεριά, από τη σκοπιά της αλληλεγγύη και από την άλλη ώστε αφορά την νόμιμη μετανάστευση μέσω της αγοράς εργασίας. Αυτή η μέθοδο είναι μεροληπτική. Και το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας δεν λύνει αυτή την ανισορροπία. Αντίθετα μάλλον. Ε, μιλάει για ηλεγγύη, αλλά προσθέτει ορισμένα φλού πράγματα και έννοιες να υποστηριχθούν τα άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Δεν πρόκειται αυτού. Κάθε άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει τα δικαιώματα που έχουμε εγγυηθεί. Και θα ήθελα αυτή η προσέγγιση να φαίνεται μέσα στο κείμενό μας ως αίτημα προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και αυτό το τμήμα το υποτιμούμε πάρα πολύ στο ψήφισμα που μας προτείνεται. Παραδείγματο χάρη, η πρόκληση που ο καθένας αναγνωρίζει. Πόσες παρεμβάσεις, πόσα ψηφίσματα, πόσες πολιτικοί λόγοι για το θέμα αυτό έξι μόνο άρθρα σε ένα κείμενο 46 άρθρων, δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν είμαστε στο ύψος της ευθύνη μας. Δηλαδή οι νομοθετικές πρωτοβουλίες να μην είναι το πολύ πολύ συμβατές με τις διεθνείς προδιαγραφές πρέπει πραγματικά 100% να συμφωνούν με τα θεμελιώδη δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που δεν είναι πολίτες αλλά που ζουν στην Ένωση. Πρόεδρος, ο κύριος Έγκστρομ. Απόν, η κυρία Μπελιέ δεν θέλει. Kalitz, Mr. Kalitz. Ο κύριος Κάλιτς, Πολωνία. Ε, ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι Ρίτσαρτ Κάλις. Είμαι ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής Δικαιοσύνης ε, του Κοινοβουλίου της ε, Πολωνίας. Χαίρομαι που συμμετέχουν και εθνικοί βουλευτές ε, στη συζήτηση για αυτό το ψήφισμα. Και ε, θέλω, θέλω να μιλήσω σε αυτό τη συζήτηση και να παρέμβω διότι ήμουν υπουργό Εσωτερικών της Πολωνίας και όταν εισήλθε η Πολωνία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα στο κοινοβουλίο μας ε, γνωρίζουμε το πρόγραμμα της Χάγης, αλλά ε, για να πούμε την αλήθεια, η εφαρμογή των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέχρι στιγμής ε, δεν ήταν πολύ ικανοποιητική. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα. Λέμε ναι, εδώ έχουμε το πρόγραμμα της Στοκόλμης για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Και απλώς επαναλαμβάνουμε το ίδιο μήνυμα. Ε, βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Πολωνία και θα πρέπει να συνδυάζεται με ολόκληρο το πρόγραμμα για την Ανατολή διότι ε, τα ανατολικά σύνορα της ε, ε, Πολωνίας είναι στη Λευκορωσία. Έχουμε 100 χιλιόμετρα από την Βαρσοβία μέχρι τα σύνορα και από την άλλη πλευρά υπάρχει δικτατορία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο για τον λαό της Λευκορωσίας να έρθει στην Πολωνία διότι χρειάζονται βίζα, θεώρηση. Οπότε όσον αφορά τις ε, ε, υπηρεσίες ασφαλείας ε, και πληροφοριών έχουμε τη Europol, την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αρχές οι οποίες καταπολεμούν τα εγκλήματα χρησιμοποιώντας όμως μυστικές μεθόδους και αυτές οι μυστικές μέθοδοι όπως τη γνωρίζουμε οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κανένα από τα κράτη-μέλη, εκτός ίσως από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν τρόπο να γνωρίζουν πού υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία μέθοδο, χρειαζόμαστε έναν τρόπο ο οποίος θα μας επιτρέψει να σηκώσουμε εκ των υστέρων τον πέπλο της μυστικότητας, δηλαδή θα πρέπει εκ των υστέρων να μπορούμε εμψυχρό να εξετάσουμε μία περίπτωση, να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν παραβιαστεί. Αυτό θα ήταν αποτρεπτικό ε, για τους ε, ε, υπευθύνους των μυστικών υπηρεσιών και θα τους αποτρέψει από το να <clears throat> παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο θέμα είναι θέμα υπηκότητος. Διότι θα έπρεπε να ενοποιήσουμε τις αρχές βάση των οποίων αναγνωρίζονται τα πολιτικά δικαιώματα στις άλλες χώρες. Ελπίζουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο με την συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε μία πρόοδο και ε, εμείς ε, έχουμε ήδη ε, κυρώσει, απλούστατα πρέπει να υπογράψουμε το προεδρικό διάταγμα και θα έχουμε έτσι σαν Πολωνή και Ευρωπαϊκή υπηκότητα πλέον της Πολωνικής. Αλλά βλέπω ότι ξεπέρασε το χρόνο μου και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Για τρία λεπτά ο κύριος Δίαφ Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαιρετώ τους τρεις προέδρους, Λόπες Αγγελάρ, Κασίνη και Μπελιγκουέρ. Επίσης, χαίρομαι για την ευτυχή εφαρμογή του άρθρου 51 του κανονισμού και να το ξανακάνουμε. Ευχαριστώ. Πολλά είναι τα επιτεύγματα της ε, διαδικασίας ε, της Χάγης, πρώην Τάμπερε. Έχουμε κάνει πρόοδους στα 10 χρόνια. Και ε, τώρα για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχουμε μεγάλες προκλήσεις και 4 χρόνια για να τις ξεπεράσουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες από αυτές. Και τώρα, επίσης έχουμε και ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί και όχι απλώς του συμβουλεύονται κάποιοι και μόνο στον προϋπολογισμό έχει πραγματική εξουσία. Θα γίνουμε κανονικό κοινοβούλιο επιτέλους. Ε, θα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα, κάποιες προκλήσεις και θα πρέπει περισσότερο να επιμείνουμε και στο αστικό δίκαιο, όπως είπε ο συνάδελφος Μπερλιγκούι, ε, αλλά και να προχωρήσουμε, και ξέρω ότι δεν είναι το ίδιο, το είπε και η συνάδελφος από το ε, Bundestag, στην ποινική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το ευρώ. Το ευρώ είναι το κοινό μας νόμισμα, αλλά είναι και ένα εργαλείο πολιτικής και οικονομικής συνοχής. Αν θέλετε είναι η κοινή μας γλώσσα και θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Και θα κάνω επικοδομητικά τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Για το κυβερνοέγκλημα, επίσης ε, σημαντικό, πρέπει να το δούμε στη Στοχόλμη, στην τρομοκρατία. Είμαστε πολύ καλοί στην καταστολή και ε, πολύ κακοί στην πρόληψη. Το 2007 ε, είχαμε 600 ε, περίπου τρομοκρατικές ενέργειες που δεν τις προλάβαμε. Ε, Eurojust, Eurojust και άλλοι τέτοιοι οργανισμοί να προχωρήσουν αλλά με κοινοβουλευτικό έλεγχο. Συμφωνώ με τον πρόεδρο Κασίνη. Να ξεπεράσουμε την κοινή μας προσπάθεια στην πρόληψη σε θέματα της μετανάστευσης και του ασύλου. Να προχωρήσουμε προς μια κοινή πολιτική επιτέλους και χρειάζεται μια πολιτική, κοινή πολιτική συγκεκριμένη και αποτελεσματική κατά της λάθρομετανάστευσης. Εννέα εκατομμύρια έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λαθρομετανάστες και θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό βέβαια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε να έρθει ο Frontex. Δεν γίνεται αυτό. Ε, τα κράτη-μέλη οφείλουν να το κάνουν με τη ε, βοήθεια και τη συνεπικούρηση της Frontex και ε, διεθνής προστασία, δηλαδή ένα καλό σύστημα ασύλου, καλύτερη κατανομή και πάρα πάρα πολύ μεγάλη ελληνική. Περισσότερη και καλύτερη προστασία των δεδομένων. Δεν χωρά καμία αμφιβολία για την ιδιωτική ζωή. Πολύ περισσότερο προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όσο έχουμε περισσότερες ελευθερίες, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε, επιγραμματικά που ξεπέρασα και το χρόνο μου. Θα κάνω επικοδομητικέ τροπολογίε μέχρι τι 22. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Yes. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζέντη. Σαρτζέντη. Not in the hall. Okay. Μάλιστα. Μάκοβεϊ, τρία λεπτά. Thank you, Chairman. Uh... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους, αν δεν ξέρουν, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια δημόσια διαβούλευση με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ερωτήθησαν 40 ερωτήσεις. Μία ερώτηση έλεγε κατά λέξη. Θεωρείτε ότι η Ένωση θα πρέπει να δώσει σε όλου του πολίτες ένα βασικό σύνολο δικαιωμάτων όσον αφορά θέματα ε, ποινικών ανακρίσεων, εγκληματικών ανακρίσεων, το 85% απάντησε ναι. Και αναφερόμαστε ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο συντάχθηκε σήμερα. Δηλαδή, όπως βλέπετε, είναι προτεραιότητα για μας και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πολιτών. Ένα άλλο θέμα και πάλι επαναλαμβάνω, εάν ε, ε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι παραπάνω για να καταπολεμήσει την διαφθορά και 88% είπαν ότι ε, ναι. Και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό που επιτύχαμε σε ένα ερωτηματολόγιο 40 ερωτήσεων. Δεν βλέπω όμως να περιλαμβάνεται αυτή η μνήα στο πρώτο σχέδιο της, ε, ε, του ψηφίσματος και γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το κοινοβούλιο θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς το λαό ότι στηρίζει τη διαφάνεια, την ακαιρεότητα στα κράτη-μέλη, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στις τρίτες χώρες και ότι στηρίζουμε επίσης και τις πολιτικές εναντίον της ε, διαφθοράς ε, σε όλες τις χώρες. Αυτή είναι η στόχη μας, να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία τέτοια αναφορά εις ε, το σχέδιο της, του ψηφίσματος και θα υποβάλω τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα όταν έχουμε ένα τέτοιο έγγραφο σαν ε, ε, το ε, έγγραφο της Στοχόλμης είναι ότι επειδή αναφέρεται σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι σαφές. Η ισχύ για τα κράτη-μέλη και για να μπορέσουμε να το τελειοποιήσουμε θα χρειαστούμε χρόνια. Αλλά φτάνει ένα, μία ματιά για να δούμε ότι ε, ε, τα βασικά υπάρχουν. Καταρχήν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ε, σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπόλ δεν υπήρξε στην Ευρώπη καμία επίθεση Ισλαμική με ε, τρομοκρατικά στοιχεία παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μας απασχολεί η Ισλαμική τρομοκρατία. Αυτό μπορεί να έρθει από εκτός της ενώσεως και ε, εκεί συμβαίνουν πολλά. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο επί του οποίου να επικεντρώνεται το πρόγραμμα. Θα μπορούσε ίσως παραδείγματο χάρη να γνωρίζουμε τι θέλει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, πράγμα το οποίο έκανε το πρόγραμμα της του Τάμπερε, το πρόγραμμα της Χάγης, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη. Οπότε θα έπρεπε εδώ να γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος στόχος μας. Όλοι θέλουμε ελευθερία και ασφάλεια, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό μήνυμα το οποίο επιζητούμε. Τι, τι λείπει. Παραδείγματος χάρη, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρακολούθηση, monitoring και η αξιολόγηση, evaluation, διότι νομίζω ότι παρόλο που τα έχουμε αναφέρει στο παρελθόν δεν έχουν επιτευχθεί. Το 2005 είχαμε μία έκθεση και βλέπουμε ότι τέσσερα χρόνια μετά στέλνεται ένα ερωτηματολόγιο στα κράτη-μέλη για να ε, ε, ε, για να απαντήσουν στο τι γίνεται με την καταγραφή των δεδομένων και είμαι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Βλέπετε λοιπόν ό,τι γίνεται θα πρέπει να εφαρμόζεται και κάπως ταχαίως. Και τέλος θα ήμουν ευτυχής αν εμείς εδώ μπορούσαμε εφόσον είναι η πρώτη κοινή συνεδρία στην οποία έχουμε τουλάχιστον στη Νέα Θητεία να δούμε πόσο μπορούν ε, να αναπτυχθούν μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέραν ε, της συνθήκης της Λισαβόνας διότι οι οκτώ εβδομάδες ε, ελέγχου για τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι ρεαλιστική προθεσμία αν γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα Εθνικά Κοινοβούρια. Οπότε θα ήταν καλύτερο να έχουμε έναν βελτιωμένο μηχανισμό να συναντιόμαστε και πιο συχνά και τέλος το πρόβλημα με τέτοια προγράμματα όπως το Τάμπερε, η Χάγη ε, και βλέπουμε ότι στη Χάγη υπάρχουν θέματα που αναφέρονται και εδώ αλλά πρέπει να μπορέσουμε να κλείσουμε τα κενά που υπάρχουν στα προγράμματα αυτά διαφορετικά ε, θεωρούμε ότι αυτονόητα θα καλυφθεί. Ο κύριος Πρόντς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε παραπάνω από ένα νομικά συστήματα. Αλλά στην Αγγλία και την Ουαλία υπάρχει μια παράδοση τεσσάρων αιώνων. Με νομολογία σταδιακά με περιπτώσεις. Άρα με φρίγη θα ακούσουν οι Άγγλοι και οι Ουαλίοι τις προτάσεις για ένα ε, ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Επίσης φρίκη είναι να αντικατασταθεί το σύστημα που έχουμε με ένα νέο σύστημα. Ω αυτά τα δικαιώματα τώρα, η επέκταση των δικαιωμάτων είναι κάτι θετικό, αλλά η δημιουργία, το έγκλημα της σκέψης τύπου όργολ και διάφορες φοβίες δεν επεκτείνουν τα δικαιώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο καταστολής και επίθεσης κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Δημοκρατική συζήτηση για την πολιτική και τη μετανάστευση πρέπει να γίνει, γιατί αυτή η πολιτική που έχουμε δεν στηρίζεται στις εμπειρίες των ανθρώπων, είτε από το ένα άκρο είτε από το άλλο άκρο. Δηλαδή, αν ακούσουμε τις εμπειρίες ανθρώπων που πλήττονται ιδιαίτερα από τη μετανάστευση, σε χώρες που, τις φεύγουν μετανάστες και χώρες που παίρνουν μετανάστες. Συνήθως που στις χώρες που λαμβάνουν τους μετανάστες είναι οι πιο φτωχοί, οι πιο ευπαθείς ομάδες που ζουν σε γειτονιές όπου υπάρχουν προβλήματα, όπου υπάρχουν κοινωνικές εντάσεις, λόγω της παρουσίας αδικαιολόγητης, λόγω της μετανάστευση και τα προβλήματα που δημιουργεί η προσπάθεια καταστολής της και ίσως αυτό που θα σα πω ίσως να μην είναι ε, να ακούσουμε και οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες που στέλνουν τους μετανάστες. Εκεί, ομάδες γυναικών, ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο, ποια είναι η γνώμη τους για το status quo της μετανάστευσης σήμερα. Είναι ικανοποιημένοι όπως εμεί νομίζουμε ότι είναι από το γεγονός ότι υποχρώνονται από γενικές οικονομικές ανισότητες και αδικίες να αφήσουν την πατρίδα τους, την οικογένειά τους πολλές την παράδοσή τους και να πάνε αλλού, διότι το, status quo μια στάση απέναντι στη μετανάστευση είναι άδικο. Άδικο. Γιατί, διότι με βάση αυτό το status quo υπάρχουν δύο κατηγορίες χωρών. Οι πλούσιες χώρες και οι φτωχές χώρες. Οι φτωχές χώρες έχουν και τις εντός αγωγικών αναπτυσσόμενες χώρες, άρα κατά κάποιο τρόπο στην Ένωση η χώρα μου η Ουγγαρία και με άλλες νέε χώρες μέλη συμβαίνει να είναι μια α, χώρα όπου ανήκει στι αναπτυσσόμενε χώρε κατά κάποιο τρόπο με βάση το διεθνέ Δομισματικό Ταμείο και οι πολίτε των φτωχών χωρών για να επιζήσουν πρέπει να αφήσουν του αγαπημένου, τα αγαπημένα του πρόσωπα εκεί που ζήσανε, τι οικογένειέ του, τι πατρίδε του και να φύγουν στι πλούσιε χώρε για να επιζήσουν. Αυτό το θεωρώ απόλυτα άδικο και θα πρέπει να δούμε σε βάθος το πρόβλημα της μετανάστευσης και να διαρωτηθούμε μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε τις ε, πολιτικές του ΠΟΕ, της Διεθνούς Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού και της Ένωση, η οποία δημιουργεί αυτή τη φτώχεια και αυτές τι αδικίες που είναι στη ρίζα του φαινομένου τη μετανάστευση. και μήπω θα έπρεπε να είμαστε υπέρ του θεμελιώδου δικαιώματο για τον άνθρωπο να μπορεί να μείνει στην πατρίδα του, στην κοινότητα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε και για να μην κινείται μόνο με αποφάσεις που διέπονται από τη λογική του κέρδους και του χρήματος και να σκεφτούμε περισσότερο με βάση την κοινότητα για ένα προσέγγιση που θα είναι και οικονομικά πιο αποδοτική αλλά ταυτόχρονα και πιο δίκαιη. Να ξαναδούμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Όλο το θέμα της μετανάστευσης να το κάνουμε συζητώντας με πραγματικούς ανθρώπους που πραγματικά ε, η μετανάστευση έχει επίπτωση στη ζωή τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μέντες Δεβίγκο, τελευταίο για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, λιγότερο θα μιλήσω. Ζήτησα το λόγο γιατί άκουσα τον κύριο Άλβαρο. Ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε. Κυρίως ένα σημείο. Το είχα σκεφτεί κι εγώ. Περνώντας όλους αυτούς τους δεδαλώδεις διαδρόμους και ατελείωτους για να έρθω εδώ. Αυτό το έγγραφο είναι πολύ ωραίο, θαυμάσιο, έχει 40 τόσες παραγράφους. Αλλά σε ένα τέτοιο θέμα έχει θεμελιώδη σημασία η επικοινωνία. Αν έρθει κάποιο να με ρωτήσει, α πούμε, περί τίνο πρόκειται το πρόγραμμα στο Χόλμη, ε, δεν έχω μία πρόταση για να εξηγήσω στο μέσο πολίτη που δεν είναι εμπειρογνώμων όπω όλοι εσεί περί τίνο πρόκειται. Και αυτή είναι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε εμείς. Μέγα τμήμα της επιτυχίας ε, του ε, σχεδίου Ντελόρ και της ενιαίας αγοράς ε, ήταν ότι όλοι ξέραμε ποιες είναι οι τέσσερις ελευθερίες. Και είχαμε μία πρόταση και τα λέγαμε. Και έλεγε ο κόσμος, α, ωραίο είναι αυτό, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών, των αγαθών και των κεφαλαίων. Λέω, με προκάλεσε ο κύριος Άλβαρα για να μιλήσω. Θα πρέπει λίγο να στύψουμε το μυαλό μας και να προσπαθήσουμε να βρούμε για τροπολογίες μία φράση, δύο, για να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε και αυτό που έχει σημασία για τον πολίτη με το πρόγραμμα της Στοχόλμης Για τα εθνικά κοινοβούλια επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό να συμμετέχουν. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, το ξέρουμε ποιο είναι. Ε, λίγο να κάνουν δουλειά και τα εθνικά κοινοβούλια, ότι είναι λίγος ο καιρός και λίγες εβδομάδες. Και για να λάβουμε σοβαρά υπόψη την πρόταση του κυρίου Άλβαρο, μια που είμαστε και παραμονές αναθεώρησης του κανονισμού, θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτή την ιδέα συνεργασίας κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εκείνε των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και προτείνω να το κάνω αυτό, να προτείνουμε ένα νέο άρθρο στον κανονισμό. Ευχαριστώ κύριε Μέντε Δεφίγου. Νομίζω σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλο του πρώτου σημείου αυτού τη ημερησία διάταξη. Και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε τους τρεις ε, εισηγητές που συνεργαστήκαμε για να κάνουμε το κοινό μας ψήφισμα. Αφού άκουσα λοιπόν όλες τις παρεμβάσεις σας, θα ήθελα να ε, σας πω τα εξή τρία. Πρώτον, αυτό το ευτυχές πείραμα της εφαρμογής του άρθρου 51 του κανονισμού μας. Δεν θα είναι η τελευταία φορά. Έχουμε χρονοδιάγραμμα εργασιών κοινή πορείας άμεσα. Στις 12 Νοεμβρίου θα ξανασυνεδριάσουμε για να ε, ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα αφού εξετάσουμε τις τροπολογίες. Στις 16 και 17 Νοεμβρίου επίσης με τα Εθνικά Κοινοβούλια ξανά και τέλος θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια βεβαίως το ψήφισμα αυτό στο Στρασβούργο στις 23 Νοεμβρίου. Αλλά εκτός από όλα αυτά την προσοχή μας συγκεντρώνει η τεράστια σημασία του προγράμματος της Στοκχόλμης εν ώψη της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ένα πολύ βασικό θέμα που είναι η ανάδειξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και ε, κατά συνέπεια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Ρωτούσε ο κύριος ε, Μέντες Δεβίγο πώς μπορούμε να συνοψίσουμε το πρόγραμμα της Στοχόλμης σίγουρα όποια και αν είναι η φράση που θα αποκρισταλώνει το πνεύμα της συζήτηση αυτή θα πρέπει να εμπεριέχει τις λέξεις δικαιώματα και πολίτες. Διότι περί αυτών πρόκειται και αυτό συζητούμε. Γι' αυτό το πρόγραμμα της Οχόλμης έχει ένα τεράστιο δυναμικό. Τονίζει τη νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης στα μάτια των πολιτών που εμείς εκπροσωπούμε. Όταν μιλούμε για ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους και να τους παρέχουμε περισσότερη ασφάλεια. Γι' αυτό και οι τρεις εισηγητές πάντα φροντίζαμε και επαγρυπνούσαμε ακριβώς για να διασφαλίσετε αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ε, ελευθερία και την ασφάλεια. Είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία να τηρηθεί και ήταν στο μυαλό μας κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά είναι σαφές επίσης ότι η ισορροπία αυτή θα απαιτήσει πολύ περισσότερη δράση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή στεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Διότι, για αρχή, σημαίνει ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο κανένα άλλο θεσμικό όργανο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και επίση ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβάλει προσπάθεια το Κοινοβούλιο για έναν εξευρωπαϊσμό, δηλαδή μεταφορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον αυτής της προσπάθειας και μεγαλύτερη προστασία από τις απειλές για τις ελευθερίες. Δεν προέρχονται αυτέ μόνο από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα οι απειλέ, αλλά και από την απώλεια της προσοχής μας, αν χαλαρώσουμε δηλαδή, αν δεν την έχουμε ε, πάντα στο μυαλό μας τόσο παρούσα. Θα πρέπει πάντα να φροντίζουμε ε, ομοιογενός και προοδευτικός να έχουμε έναν ανταγωνισμό προς τα πάνω και όχι μια κούρσα προς τα κάτω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Από πλευράς μεθόδου τώρα και ο Λουίτζι Μπελεγκουέλ και ο Κάλλος Κασίνη και εγώ σημειώσαμε αυτό που μας είπατε, ότι θα κάνετε τροπολογίες μέχρι τις 22 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία και θα τις ε, υποδεχθούμε με ανοιχτό πνεύμα και πρόθυμη για συνεργασία με τις πολιτικές ομάδες, έτσι ώστε τελικά να έχουν και νόημα οι τροπολογίες. La, la... Τελικά ε, θα ήθελα να σας πω ότι το κείμενο που σας μοιράσαμε σήμερα ε, είναι η τελευταία εκδοχή. Υπήρχαν και προηγούμενες. Η πρώτη, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ πιο μακροσκελής. Και σιγά σιγά μετά από τις συνεδριάσεις που κάναμε και τη συνεργασία, περιορίστηκε το κείμενο. Συρρυκνωνόταν κάθε φορά, ήταν και πιο συνεκτικό. Γι' αυτό πολλές ειδικέ αναφορές για να συνεργαστούμε σε ε, ε, με τις τρίτες χώρες προέλευσης των μεταναστών κτλ για να διορθώσουμε τις αδικίες που βρίσκονται στη ρίζα της λαθρομετανάστευσης ή της μετανάστευσης. Σιγά σιγά, επειδή συμπυκνώθηκαν αυτές οι ιδέες, έχουν χάσει έτσι, εκφραστικότητα θα έλεγα. Δεν είναι πολύ αναλυτικές οι ε, περιγραφές και για τα θύματα. Δηλαδή κάθε παράγραφος με την πάροδο του χρόνου περιοριζόταν σε μέγεθος, άρα και ήταν και πιο συμπυκνωμένη η περιγραφή των ιδεών. Δεν είναι ότι λείπουν. Πάντως ε, οι τροπολογίες θα μας βοηθήσουν για να ξαναπούν πολλά από αυτά τα σημεία ε, όπως θέλετε. Τέλος, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό που δύσκολα καταλαβαίνουν και αισθάνονται οι πολίτες που είναι αυτά τα κανονιστικά εργαλεία που έχουμε από τον πρώτο πυλώνα και τον τρίτο πυλώνα, αυτή η ιστορία σιγά σιγά θα λήξει. Έχει ημερομηνία λήξη. Στη χειρότερη περίπτωση πέντε χρόνια. Πάντω είναι μετρημένες οι μέρε του. Είναι λίγα τα ψωμιά του. Από εδώ και πέρα όλο αυτό το κοινοτικό εκτιμένο οι αποφάσεις πλαίσιο, οι μεγάλες πρόοδοι που έχουν γίνει, περιέχουν ένα τεράστιο δυναμικό συμμετοχής και νομιμοποίησης για να καταλαβαίνει και ο πολίτης ότι αυτά που κάνουμε έχουν νόημα για να βελτιώσουν τη ζωή του, ναι, για περισσότερη ελευθερία και περισσότερη ασφάλεια. Όλα αυτά θα γίνουν σε ένα πολύ άμεσο μέλλον. Ότι θα έχουμε περισσότερη Ευρώπη και ε, οφείλουμε αυτό να το μεταδώσουμε και στους πολίτες. Θα ακούσουμε τώρα τον Κάρλο Καζίνη και τον Λουίτζι Μπελιγουέν, αλλά ας μην ξεχάσουμε ότι πριν τελειώσουμε έχουμε και ένα θέμα και για τις τροπολογίες αλλά και τις προφορικές ερωτήσεις. Δύο τον αριθμό που θέλω να πω κάτι τελευταίο τι θα κάνουμε με αυτά. Τα έχετε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτό που είπατε εσείς. Ας περιμένουμε τις τροπολογίες, να τις ενσωματώσουμε στο κείμενο, να το βελτιώσουμε. Προσωπικά με παραξένεψε από μερικές παρατηρήσεις που άκουσα. Πρώτα, το πόσο σημαντικό είναι το αστικό δίκαιο. Για το ποινικό δίκαιο ακούσαμε ότι είναι δύσκολο να το εναρμονίσουμε. ιδιαίτερα όσον αφορά τον δικαίωμα από την πλευρά του συνηγόρου, αλλά για το ποινικό δίκαιο, ενδεχομένως η συνθήκη της Λισαβόνας να μας επιτρέψει να έχουμε διασυνοριακά αδικήματα. Δεν ξέρω, πέραν αυτού δεν μπορούμε να πάμε. Αντίθετα για το αστικό δίκαιο, οι πολίτες που έχουν παρεδώσει με επιχειρήσεις που έχουν που λειτουργούν σε πολλές χώρες ταυτόχρονα θα είναι πιο εύκολο, πιο εύκολη από εδώ και μπρο η πρόσβαση στη χρήση αυτού του δικαίου. Σωστά κάποιος τόνισε επίσης ότι στο κέντρο πρέπει να είναι ο πολίτης αλλά και ο άνθρωπος. Συμφωνώ επίσης με μια άλλη υπογράμμιση όσον αφορά την ασφάλεια και τη σύνδεσή της με την μετανάστευση. Ασφάλεια φυσικά σημαίνει να καταπολεμείται το οργανωμένο έγκλημα. Ιδιαίτερα όταν εκμεταλλεύεται ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν πρόσφυγες από τη βία, από τον πόλεμο, από την πείνα και πέφτουν στο οργανωμένο έγκλημα και τα δίχτυα του. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμούνται αυτού του είδους οι οργανώσεις. Βέβαια είναι τέτοιο κείμενο, δεν μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες. Μοιραία είναι γενικό. Το πρόγραμμα περαιτέρω πρέπει να εκπονείται χρόνο με το χρόνο με λεπτομέρειες. Σημειώσαμε τις παρατηρήσεις σας και εμείς υπεύθυνοι από την πλευρά της Επιτροπής συμφωνούμε με αυτά που υπόθηκαν και ο κύριος Μπερλιγκουέρ προσθέτω σε αυτά που είπε ο Κάρλο Καζίνη. Παρακαλούμε αυτούς που έκαναν τις παρατηρήσεις να κάνουν τροπολογίες. Αυτό θα μας διευκολύνει. Πολλά από όσα υπόθηκαν με έπεισαν ότι πρέπει τα στοιχεία αυτά να μπουν στο κείμενο. χωρίς φυσικά να το κάνουμε πολύ μακροσκελές το κείμενο. Στις 22 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι λύγει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Τρεις σκέψεις. Η μία, κάποιος είπε ότι τα εθνικά νομικά συστήματα δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε σε αυτά, γιατί έχουμε την Ευρώπη των κρατών. Ναι, αλλά στην Ευρώπη πρέπει να συμβιώσουμε με τα εθνικά προγράμματα. Και οι πολίτες μετακινούνται, οι επιχειρήσεις μετακινούνται. Με παραξένεψε πολύ από την η εμπειρία μου. Η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα ότι στην Αγγλία, την Ουλία, τη Σκοτία και τη Βόρεια Ιρλανδία, τελείως διαφορετικά συστήματα. Είναι σαν να λέμε η Λουιζιάννα, ας πούμε, δεν συμφωνεί με τα άλλα κρατήδια στι ΗΠΑ. Πολιτείες. Συμβιώνουμε στα κράτη μας. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος μέσω μιας διαδικασίας. Κανένας δεν θέλει να κάνει νόμους που να πέφτουν από πάνω. Κραπ. Τη διαδικασία αυτή την ζητάει η κοινωνία. Οι πολίτε που μετακινούνται θέλουν να έχουν την βεβαιότητα του δικαίου σε άλλο κράτος μέλος. Αν πάνε. Το θέλουν αυτό. Το ζητάνε. Οι επιχειρήσεις θέλουν βεβαιότητα δικαίου. Να μπορούν να επιλύσουν τις διάφορες διαφορές που έχουν είτε με μεσολάβηση είτε προστρέχοντας, προσφεύγοντας σε ένα δικαστήριο. Έχουν και αυτές την ανάγκη να μετακινούνται, μετακινούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σέγγεν. Πιστεύω λοιπόν ότι τα κοινά βήματα θα οδηγήσουν σε προσέγγιση των συστημάτων στην Ένωση η ριζική διαφορά μεταξύ common law και civil law του κρατού και του άγραφου δικαίου έχει μειωθεί. Υπάρχει από τη μια μεριά μια νομολογία των δικαστηρίων. Εμείς στην υπηρετική Ευρώπη με το, νομικό, το ρωμαϊκό δίκαιο κλπ. Είχαμε διαφορετικό σύστημα. Αυτή όμως είναι η δύναμη, η δύναμη της δικαστικής νομολογία. Σήμερα όμως έχω μια κοινωνία της ταχύτητας, όχι κωδίκων που μένουν χωρίς την παραμικρή αλλαγή επί αιώνες. Είμαι καθηγητής κωδικοποιημένου δικαίου και σας τα λέω παρόλα αυτά, σας τα λέω αυτά. Αυτή είναι η κοινωνία σήμερα. Ένα άλλο παράδειγμα. Το δικαίωμα του στο δίκαιο των συμβάσεων. Αν μετά από 27 δίκαια συμβάσεων βγει ένα πλαίσιο κοινή αναφοράς, διαγράφεται από πίσω, ότι μπορούμε να επιλέξουμε το ένα και όχι το άλλο. Αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλο δίκιο. Το πλαίσιο αναφοράς, το κοινό πλαίσιο αναφοράς, αυτό θα επιτρέψει στον και στην επιχείρηση να βρει το δρόμο του. Η εσωτερική κινητικότητα και η εσωτερική διαδικασία αυτή ακριβώς είναι. Για το διαζύγιο Υπάρχουν πτυχέ του οικογενειακού δικαίου που επιβάλλονται σήμερα. Υπάρχουν διαφορετικέ κουλτούρε βέβαια που συμβιώνουν σήμερα, νομικέ εννοώ. Που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση. Evaluation σημαίνει δύο πράγματα. Παρακολούθηση και αξιολόγηση. Παρακολούθηση καταρχήν, εποπτεία τη διαδικασία αυτή. αυτό απαιτείται, διαχρονικά. Και μετά αξιολόγηση, να δούμε τα αποτελέσματα. Και αυτό χρειάζεται. Ευρωπαϊκή νομική κουλτούρα. Αυτό υπάρχει στη βάση όλων αυτών. Το ζητάμε από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο επένδυση στην κουλτούρα, διότι η κουλτούρα αποδίδει, δίνει αποτελέσματα, παρέχει όφελος, γνώσεις, εμπειρία, μαθητεία, όλα αυτά είναι μέσα στο, στην έννοια αυτή της κουλτούρας που ανάφερα. Άλλο ένα από την εμπειρία μου, γιατί προείδρευσε ενός δικτύου, ευρωπαϊκού δικτύου, για συμβούλους στους δικαστές. Και ασχολήθηκα με τον κοινό αυτό χώρο, από τη σκοπιά, με τα μάτια της δικαιοσύνης. Ε, λοιπόν, υπάρχουν 7 περίπου δίκτυα των οτάτων δικαστηρίων, εισαγγελέων κλπ. στην Ευρώπη. Υπάρχει και ένα δίκτυο για την κατάρτιση δικαστών. Ε, λοιπόν, η Ευρώπη απαρτίζεται από θεσμικά άργωνα από προδιαγραφές και από μορφές συνεργασίας ενδοκρατικές. Αν καταφέρουμε να έχουμε επαφή με αυτές τις δομές που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δικηγόρους κλπ, θα συνοδεύσουμε την θεσμική πρωτοβουλία που χρειάζεται αλλά δεν αρκεί, με αυτούς που είναι το δίκτυο της παρουσίας των φορέων της δικαιοσύνης. Ζητάμε δηλαδή να βοηθήσει η Κομισιόν και το Συμβούλιο αυτή η προσπάθεια που θα έρχεται από κάτω, που προωθείται από κάτω, να βοηθηθεί συγκεκριμένα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Το τελευταίο σημείο της κοινή αυτής συνεδρίασης έχουμε την τυπική έγκριση της προθεσμίας για τροπολογίας 22 Οκτωβρίου συμφωνούμε και η έγκριση δύο προφορικών ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν ερώτηση προς το Συμβούλιο έχει, σας έχει μοιραστεί αναφέρεται στη σημασία της δράσης έτσι ώστε η μεταφορά όλων αυτών των κεκτημένων τρίτου πυλώνα στο ευρωπαϊκό δίκαιο στο προσεχές μέλλον και η ερώτηση προς την Κομισιόν σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουν μοιραστεί οι ερωτήσεις. Έχουν διανεμηθεί. Ο κύριος Νταφ Έχουμε μόνο την ερώτηση προς την Κομισιόν. Μόνο αυτή διανεμήθη, τουλάχιστον σε μένα. Πρόεδρος, θα πρέπει να υπάρχει και η... άλλο ένα φύλλο. Υπάρχει, αν θέλετε μπορείτε να το πάρετε, η ερώτηση προς το Συμβούλιο. Σας τη διαβάζω. Τι λέει. Τι δράση θα αναλάβει το Συμβούλιο θα φορά στο χώρο ελευθερία ασφάλεια και δικαιοσύνη για τα επόμενα πέντε χρόνια, λαμβάνοντα υπόψη το ότι όταν θα ισχύσει η συνθήκη τη Λισαβόνας, η Ένωση θα δράσει στι περισσότερες περιπτώσεις με βάση την τακτική νομοθετική διαδικασία. Και άλλη ερώτηση. Τι δράση σκοπεύει να λάβει συγκεκριμένα προκειμένου να επικαιροποιήσει και να προσαρμόσει το κεκτημένο σύμφωνα με τη νέα θεσμική κατάσταση. Αυτή είναι η ερώτηση προς το Συμβούλιο. Θα σας διαβάσω και την ερώτηση προς την Κομισιόν. Όταν η Κομισιόν υποβάλλει τις προτάσεις της προκειμένου να ευθυγραμμιστεί τα κεκτημένα με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα φροντίσει να δοθεί δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετέχουν με βάση προτάσεις που θα έχουν αναθεωρηθεί και όσον αφορά τη διαδικασία και όσον αφορά την ουσία. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Θα σταλούν οι ερωτήσει αυτές στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Μία τελευταία λέξη εκ μέρους της Προεδρίας Συμβουλίου για να τελειώσουμε. Επειδή το πρόγραμμα της Στοχόλμη θα έχει το όνομα της πρωτεύουσα της Σουηδίας. Κύριε Νίλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα σας κρατήσω για πολύ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε επαφές στο άμεσον μέλλον. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε ένα θέμα απαντώντας στον κύριο Μέντες Ντεβίγκο Νομίζω ότι έκανε τη σωστή ερώτηση. Τι είναι το πρόγραμμα της Στοχόλμης. Κανείς δεν το έχει δει, δεν υπάρχει. Ελπίζω θα υπάρχει μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου. Αλλά από κοινού Σουηδική Προεδρία, το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, η κοινωνία των πολιτών και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν εμπλακεί θα μπορέσουν μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου να πούν ότι θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μία ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη προς όφελος των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νίλσον. Όλοι συμφωνούμε με την ελπίδα σας και ελπίζουμε ότι θα έχει υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ε, Στοχόλης μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου. Τώρα λοιπόν λύεται η συνεδρίαση μέχρι τις 12 Νοεμβρίου αυτής της κοινή Επιτροπής.